και φυσικά έχει πολλές <clears throat> επιπτώσεις για τις εμπορικές μας σχέσεις. Γιατί πολλές φορές θέτουμε εμείς σε πολλές εμπορικές συμφωνίες το θέμα της ε, ε αποτροπής χρηματοπιστωτικών ρευμάτων που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση της ε, διαφθοράς και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρούμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το χρηματοπιστωτικό τομέα πέραν της φιλελευθερωποίησης του τομέα αυτού. Και νομίζω ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο. Έχουμε ζητήσει να εκπονηθεί μία μελέτη για το θέμα αυτό. τον Απρίλιο του 2016 δημοσιεύτηκε αυτή η έκθεση και εδώ <clears throat> η συγκητής για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Μορέλ, στον οποίο δίδω ασμένος τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Μορέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Συνάδελφοι, είπατε και εσείς ότι το Κοινοβούλιο εδώ και μερικούς μήνες έχει αρχίσει να ασχολείται μετά από μια σειρά σκανδάλων με το θέμα της φοροδιαφυγής. Είναι σκάνδαλα λοιπόν τα οποία έχουν προκαλέσει έτσι αναταραχή στην κοινή γνώμη και επομένως έχει κυκλοφορήσει ε, έχουν ξεκινήσει κάποια κείμενα έτσι ώστε να ε, αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Τώρα όσον αφορά ε, την βελτιστοποίηση, την φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και το ξέπλυμα, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι περίπλοκο και γι' αυτό ακριβώς συζητούμε τώρα για ένα ειδικό κείμενο. Όπως σας είπα, ε, ε, το εμπόριο ε, υπηρεσιών, κυρίως χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό η οδηγία ε, για το ε, ξέπλυμα χρήματος και για τη χρήση του χρήματος αυτού ε, για, τη, για τρομοκρατικές ενέργειες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως το θέμα των ενδιάμεσων, των τραπεζικών και άλλων είναι κάτι που μας απασχολεί, πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό όπως είπατε. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή μας προτείνει κάποια στοιχεία έτσι ώστε να ενισχυθεί ε, και το εμπορικό αλλά και το θεσμικό ε, σκέλος ε, των, του ξεπλήματος του χρήματος. Εγώ προτείνω τα εξής. Εάν θέλουμε ε, να είμαστε αξιόπιστοι, θα πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουμε με διαφάνεια και επομένως αυτό θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό κριτήριο σε διεθνές επίπεδο και επομένως επαναλαμβάνω ε, σε μια, επαναλαμβάνω μια πρόταση που μας είχε κάνει ε, ο κύριος Στίγκλιτς, βραβείο Νόμπελ, οικονομίας και τα λοιπά, σε μια ακρόαση ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει διαφάνεια. Δεύτερον, έχουμε αργήσει ως δημόσια διοίκηση γιατί οι καινοτομίες όσον αφορά την βελτιστοποίηση και την φοροαποφυγή ε, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από μας ε, και ε, επομένως ο μόνος τρόπος ε, για να προχωρήσουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο των θετικών καταλόγων. Δηλαδή όταν σε μια εμπορική συμφωνία αναφερόμαστε σε χρηματοοικονομικά θα πρέπει να αναφερόμαστε και σε θετικές λίστες και σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μια σχετική κάλυψη όσον αφορά αυτές τις μεθόδους φοροαποφυγής. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να καταπολεμήσουμε κάποιες στρατηγικές φοροαποφυγής μέσω μεγαλύτερης επαγρύπνησης στη διάρκεια τη, στιγμή ε, της σύνοψης εμπορικών συμφωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα η Σκιώδης, όσοι είναι εδώ τουλάχιστον. Και ακολουθεί κυρία Χράντσοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γενικά εμείς χαιρετίζουμε την πρόταση της Κομισιόν η οποία θα επικαιροποιήσει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ε, έκπληση χρημάτων, χρηματοδότηση ε, τρομοκρατίας και φοροαποφύγης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και το εμπόριο είναι ένα τομέα ο οποίο εμπλέκεται σε όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή γιατί εισήγαγε και την διάσταση του εμπορίου σε αυτή την πρόταση. Έχω όμω ορισμένε και, και ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή μα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία τη για να προτείνει λύσει για το πώ μπορούμε να αναχαιτήσουμε τι παράνομε ροέ χρημάτων, πώ μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε του κινδύνου ξεπλήματος χρημάτων με επικοδομητική εμπορική πολιτική. Είναι γεγονός ότι το ελεύθερο εμπόριο μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους ξεπλήματος χρημάτων. Τα στοιχεία όμως από διάφορες μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ του ελευθέρου εμπορίου και της αύξησης των παρανόμων ροών χρημάτων. Το εμπόριο υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό των συστατικό στοιχείο τη επόμενη γενιά εμπορικών συμφωνιών, Ιδίω όταν προδίδει την τεχνολογία και την κινητικότητα των εργαζομένων. Μπορούν να υπάρχουν κάποια κενά και παραθυράκια σε ό,τι αφορά τι ε, ε, ρυθμίσεις για διαμεθοριακές υπηρεσίες, αλλά αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν ευκαιρίες οι οποίες δεν πρέπει να θυσιαστούν και είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον μακροχρόνιο χρόνο στόχο μας που είναι η πολυμερής αναπτύξη του εμπορίου. Αυτή τη στιγμή Έχουμε υποστεί σημαντικές ε, ε απώλειες από τη μην έγκριση συμφωνιών και αυτό είχε και ε, απώλειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επομένως, οι συμφωνίες δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι κίνδυνος, θα πρέπει εμείς να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας για να επιτύχουμε τους κυρίους μας στόχους. Θα πρέπει να ζητήσουμε και οι εταίροι μας εμπορικοί να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διαφάνειας, αλλά δεν θέλουμε να κόβουμε τις επαφές μας όταν δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με το ξέπλυμα χρημάτων είναι η διαφορά μεταξύ της έγκρισης νομοθεσίας και της εφαρμογής, της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας για τον έλεγχο του ξεπλήματος χρημάτων. Θα πρέπει να δώσουμε τη δική μας συνεργασία και βοήθεια για να εξασφαλίσουμε ότι τηρούνται αυτά τα πρότυπα. Η ομάδα μας θα καταθέσει και μερικές τροπολογίες και προσβλέπω και στην περαιτέρω συζήτηση για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή. Νομίζω ότι το προτινόμενο σχέδιο γνωμοδότησης πηγαίνει στην σωστή κατεύθυνση και χαιρόμαστε γι' αυτό. Βέβαια δεν πήγαμε λίγο παραπέρα, δεν το κάναμε πιο ισχυρό διότι θεωρούμε ότι το θέμα της χρηματοπιστωτικής απάτης δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο, αλλά και τις εμπορικές συμφωνίες. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε και κάποιες διατάξεις για να προλάβουμε αυτή την απάτη, ειδικά στις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ε, ας πούμε, ε, να πάμε λίγο παραπέρα από τις συνήθεις δεσμεύσεις για την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Τώρα, Κάποιες, κάποιοι ορισμοί ε, μιλάνε για του, τα μητρώα των ε, πραγματικών δικαιούχων, ε, για την, τις πολιτικές εταιρικής φορολογίας. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Νομίζω όμως ότι πάνε στην ίδια κατεύθυνση με τον εισηγητή, αλλά λίγο παραπέρα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς αν διαφωνούμε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι μόνο λοιπόν το εμπόριο όπως είπα πριν, αλλά είναι και οι εμπορικές συμφωνίες που πρέπει να θυγούν και γι' αυτό ε, έχουμε ε, πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε ε, ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να υποστηρίξω αυτή την γνωμοδότηση. Ένας από τους λόγους που υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση είναι ότι κάποιοι τομείς διαφεύγουν του ελέγχου τους ε, και ότι δεν έχει αντικατασταθεί ο έλεγχος αυτό σε άλλο επίπεδο. Η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή, η αλλαγή χεριών στα, όσον αφορά την κατοχή χρημάτων, το ξέπλυμα χρήματος, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι ζητήματα που τους απασχολούν. Ο εισηγητής λοιπόν έχει καταφέρει να πετύχει μια πολύ καλή ισορροπία στις ε, τροπολογίες. Ε, συμφωνώ με τα όσα ε, λέει ο συγητής, θεωρώ ότι ακριβώς ε, ε, αυτό πετυχαίνει ο συγητής, την ισορροπία. Οι τροπολογίες της κυρίας Κέλλερ ω πηγαίνουν πιο μακριά. θεωρώ ότι είμαστε στην καλή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στην Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Just, η Πολύ Βάιν Τσίρεν. Η κυρία Καλούμπα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Δεν έχω ιδιαίτερα σχόλια γιατί ε, η συνάδελφος από την DigiTrade ίσως ε, θα κάνει πιο λεπτομερή σχόλια, αλλά πάντως σε γενικές γραμμές να πω ότι εμείς καλοδεχόμαστε την ε, αντιμετώπιση που είχε η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το ξέπλυμα του χρήματος. Ε, όσον αφορά τον κατάλογο των ε, χωρών ε, που αναφέρει ο εισηγητής σε κάποιο σημείο της έκθεσής του, είμαστε διατεθειμένοι να δούμε από κοντά αυτό το οποίο υποβάλλεται, αλλά θα ήθελα να, ζητήσω, να σας ζητήσω να δώσετε τον λόγο στη συνάδελφό μου από την DigiTrade. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ για, τις, για την γνωμοδότηση, το προσχέδιο γνωμοδότηση και τι παρεμβάσει. Ε, υπήρξαν ανταλλαγέ απόψεων ε, και νομίζω ότι κάποιε από τι προτάσει που αναφέρθηκαν εδώ είναι πολύ θετικέ. Ε, και βεβαίω και η αναγνώριση ότι θεωρούμε όλοι ένα πολύ σημαντικό θέμα και, και αυτό είναι πολύ θετικό. Και μάλιστα και στην ανακοίνωσή μας όσον αφορά ε, το θέμα αυτό γίνεται ιδιαίτερη ε, επισήμανση για την ε, διαφθορά καθώς επίσης και για το ξέπλυμα του χρήματος και επομένως και εμείς θέλουμε να δούμε από κοντά το θέμα της ενίσχυσης των ρητρών που θα αφορούν αυτό το ζήτημα και που θα συμπεριληφθούν στις εμπορικές συμφωνίες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και αυτό που αναφέρεται και το θέμα του beneficial ownership ε, είναι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε ε, να υπογραμμίσουμε ότι είναι σημαντικό όταν μιλάμε για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να υπενθυμίσουμε ότι οι εμπορικές μας συμφωνίες συνήθως δεν συμπεριλαμβάνουν ε, δεσμεύσεις ε, που αφορούν τις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ε, συναλλαγές αλλά αναφέρονται σε εγκατεστημένους εμπορευόμενους και επομένως δεν είναι σαφές ότι υπάρχει μια τέτοια σχέση αιτίου αιτιατού αν θέλετε ανάμεσα σε εμπορικές συμφωνίες και την απελευθέρωση αυτών των κινήσεων. Εμείς εστιαζόμαστε κυρίως στο establishment στην εγκατάσταση. Κάτι άλλο το οποίο θέλουμε να υπογραμμίσουμε και το οποίο αναφέρεται εδώ είναι το ζήτημα του κατά πόσον οι απαιτήσει καλής διακυβέρνησης ε, και θέματα ε, ξεπλήματο ε, χρήματο θα πρέπει να συνδεθούν με τρόπο δεσμευτικό με τις εμπορικέ συμφωνίες. Είναι σημαντικό νομίζω να δούμε το στον συνεργατικό χαρακτήρα, δηλαδή αναφέρομαι στις αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες, οι οποίε χρειάζονται βοήθεια έτσι ώστε να αναπτύξουν τρόπου κατά καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος χρήματος. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεργατική προσέγγιση στις ε, συμφωνίες ε, συνεργασίας και οπωσδήποτε να προβλέπονται και κεφάλαια τεχνικής αρρωγής. Ήδη έχουμε στην διάθεσή μας πολλά εργαλεία και βεβαίως αναπτύσσεται και ένα νομοθετικό πλαίσιο ε, για το ξέπλυμα χρήματος. Αυτό το ανέφερε ε, και η ε, συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, G-Just. Βεβαίως υπάρχουν κατάλογοι με τις χώρες υψηλού κινδύνου και τους τομείς υψηλού κινδύνου. Πάντως έχουμε και μηχανισμούς και έχουμε μηχανισμούς και εργαλεία έχουμε ας πούμε την Financial Action Task Force ε, καθώς επίσης ε, και ομάδες ε, καταπολέμησης του ξεβλήματος χρήματος που ήδη δουλεύουν πάνω στα θέματα αυτά. Όλα αυτά σας τα είπα για να καταλήξω ότι μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα, ότι το δουλεύουμε από κοντά, ότι ήδη έχουμε βάλει κάποιες τέτοιες πτυχές και στις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και ότι θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και υπό το φως των προσφάτων εργασιών που έχουν λάβει χώρα ε, στο, στα πλαίσια του ΟΣΑ και άλλων οργανισμών. Ε, οπωσδήποτε όλοι ε, θέλουμε να προσεγγίσουμε σωστά το θέμα αυτό και έτσι άλλωστε δικαιολογείται και η πολλή δουλειά που κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αλλού. Οπωσδήποτε στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να βελτιωθεί και η καλή διακυβέρνηση η οποία θα φέρει καλά αποτελέσματα και στον τομέα των συναλλαγών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κοινή γνώμη. Είναι σημαντικό να υπάρξει έλεγχος του χρηματοπιστωτικού συστήματος που οι πολίτες του αντιλαμβάνονται εκτός ελέγχου. Έχει χαθεί μια σημαντική φορολογική ύλη που υπολογίζεται σε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την Αφρική. Βέβαια η δημιουργία ικανοτήτων στο δημόσιο μηχανισμό είναι απαραίτητη για να έχουμε ένα <clears throat> πραγματικό ελεγκτικό σύστημα. Τα 40 λοιπόν αυτά δισεκατομμύρια των Αφρικών πρέπει να πάνε στα αφρικανικά κράτη για να, να γυρίσουν στα αφρικανικά κράτη και να χρησιμοποιηθούν για δημιουργία υποδομών και παιδεία. Δίνω και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Πάρα πολύ εν συντομία, γιατί κύριε Πρόεδρε, εγώ συμμερίζομαι απόλυτα αυτό που είπατε. και εγώ πιστεύω, όπως και η Κομισιόν, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ρήτρα ευκυβερνησίας, αλλά θα πρέπει να έχει και δεσμευτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό ακριβώς εμείς ζητούμε να υπάρχει η φορολογική ερεσιμότητα στις συμφωνίες αυτές γιατί αυτό είναι ένα νέο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Κατά τα άλλα και εγώ συμμερίζω με τις απόψεις των συναδέλφων μου. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο στεναρό το, το κείμενο αυτό. Στην κυρία Σκάκελε θέλω να της πω ότι θα συζητήσουμε και τις τροπολογίες αλλά έχουμε ένα περιορισμένο χώρο σε αυτή τη γνωμοδότηση υπό την έποψη των αριθμού χαρακτήρων και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό των μητρών, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και, αμ και υποχρεωτική <clears throat> ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν για ξέπλυμα χρήματο. Δεν είναι θέμα λοιπόν έλλειψη στεναρότητα. Από μένα απλώ είναι περιορισμένο ο χώρο στη γνωμοδότηση, αλλά πιστεύω ότι μαζί με του άλλου κοιοδησίτε θα καταλήξουμε σε ένα ενδιαφέρον κείμενο το οποίο θα μπορέσει να επιτύχει μια σύνδεση μεταξύ του διεθνούς εμπορίου και της καταπολέμησης της, ε, ε, του ξεπλήματος χρήματος που ενδιαφέρει πολύ τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ πολύ και πρόεδρος. Να σας πω ότι έχουμε. Έχουμε κάπως ένα ασθενό χρονικό πλαίσιο. Η προθεσμοί για τις τροπολογίες. Εκπνέει αύριο, 30 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα, το μεσημέρι. και έχουμε αποφασίσει να εξετάσουμε αυτές τις ε, τροπολογίες στα αγγλικά. Ακόμα συνένεσε και ο γαλλόφωνος εισηγητής σε κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι δυνατό. Ε, ή αν ήταν δυνατό θα μπορούσαμε να δουλέψουμε όλοι στα γαλλικά. Αλλά επομένως όλοι έχουν δεχτεί μέχρι αύριο το μεσημέρι να κατέθουν οι τροπολογίε <clears throat> ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το ταχύτερο δυνατό τη γνωμοδότησή μα. Πάω τώρα στο σημείο 11. Εμπορική Συμφωνία <clears throat> Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Δημοκρατία της Κορέας. Εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με την Νότια Κορέα. 1η Ιουλίου του 2016 έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ε, θέση σε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Μάλλον όχι η θέση σε εφαρμογή, η προσωρινή εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Γιατί μόνο πέρσι έγινε η επίσημη εφαρμογή αυτής της ε, συμφωνίας όταν το Ιταλικό Κοινοβούλιο ως τελευταίο κοινοβούλιο κύρωσε αυτή τη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας εφαρμόζονται εδώ και πέντε χρόνια ήδη και επομένως είναι καιρός να κάνουμε μια αναθεώρηση της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, να δούμε ποια θετικά αποτέλεσματα έχουν προκύψει, ποιε είναι οι προκλήσεις και, τα, και οι δυσκολίες που συνδέονται με αυτή την συμφωνία. Για μένα είναι προφανές ότι η κατάσταση των εξαγωγών των ευρωπαϊκών προς την Κορέα έχει βελτιωθεί μέσω αυτής της συμφωνίας από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα για την εφαρμογή του κεφαλαίου βιωσιμότητος. Ώστε λοιπόν να δούμε καλύτερα τα θέματα αυτά, στείλαμε καταρχήν μια αντιπροσωπεία στη Βόρεια, στη, όχι στη Νότια Κορέα, στο πρώτο ήμιση αυτού του έτους και επίσης έχουμε και ένα μόνιμο εισαγητή, ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα αυτά, ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει πώς προχωρεί η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και με μεγάλη χαρά έχω, έχουμε την ε, παρουσία του κύριου Σάινφελτ, ο οποίος είναι ο συγητής μας και ο οποίος μπορεί να παρουσιάσει την αντίστοιχη έκθεση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. για, η οποία στην ουσία συνοψίζει με τον σύντομο αλλά πολύ αποτελεσματικό χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη συμφωνία, Έχουμε εξετάσει την εφαρμογή της ε, FTA με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νότια Κορέα και θέλουμε να δούμε αν στην ουσία, οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται στην πράξη και αν και οι στόχοι της συμφωνίας ε, επιτυγχάνονται. Τίποτα δεν είναι τέλειο βέβαια. Και τίποτα δεν μπορούμε να το πετύχουμε 100%. Φαίνεται όμως ότι η συμφωνία εφαρμόζεται θετικά, πολύ θετικά. Και τα αποτελέσματα το, της συμφωνίας, ειδικά από τη δική μας πλευρά, είναι απτά, είναι πρακτικά και συνάδουν με τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σε γενικές γραμμές ε, χαιρετίζουμε αυτή τη συμφωνία. Πριν κατατεθεί λοιπόν το σχέδιο της έκθεσης για αυτή τη συμφωνία, έγινε μια πολύ ολοκληρωμένη ανάλυση. Εξετάσαμε στατιστικά δεδομένα και άλλα στοιχεία. Ο σκοπός μας ήταν να διαπιστώσουμε την εποκατάσταση της ε, επίσημης εφαρμογής της συμφωνίας, αν υπάρχει δηλαδή αποτελεσματικότητα σε οικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο ε, σε απτούς τομείς. Ε, για παράδειγμα, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια εξέταση όλων των τομέων που είναι πιο πρακτική και είχαμε και μια υποκειμενική αξιολόγηση ε, η οποία βασίστηκε σε συναντήσεις με τους δικαιούχους και από όλες τις πλευρές. Να έχουμε λοιπόν, είχαμε επαφές όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και στη Σεούλ. Πήγαμε στην Κορέα καταρχήν, αλλά και πέρυσι το Δεκέμβρη στις Βρυξέλλες είχαμε κάποια εργαστήρια στα οποία είχαμε προσκαλέσει διαφόρους εκπροσώπους των αρχών του ιδιωτικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών θεωρώ ότι έχουμε πλέον πολύ καλή γνώση και των συγκεκριμένων, των απτών και των λιγότερο συγκεκριμένων και απτών αποτελεσμάτων της συμφωνίας. Οι δικαιούχοι είναι στην ουσία αυτή που μας έδωσαν αυτές τις πληροφορίες, μιλώντας μαζί μας. Στο πρώτο τμήμα της έκθεσης αναφέρω μια σειρά δεδομένων και στοιχείων που αναφέρονται βέβαια πολύ συνοπτικά γιατί υπάρχουν κάποιες, κάποιοι τυπικοί περιορισμοί σε σχέση με το μέγεθος αυτού του τμήματος αλλά στην ουσία αυτό το τμήμα της έκθεσης μας γνωστοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα της συμφωνίας. Στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης έχω αναφέρει επιγραμματικά μια σειρά από ζητήματα, ας πούμε μη δασμολογικούς ε, φραγμούς, ε, υγειονομικούς φραγμούς, ε, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρόσληψη της συμφωνίας από τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές. Ένα μειονέκτημα που βλέπω, το οποίο δεν έχει να κάνει με την συμφωνία αυτή καθεαυτή, αλλά με τις σχέσεις μας, είναι ότι μάλλον θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα στο επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συμφωνία περισσότερο προς όφελός τους. Όμως αυτό έχει να κάνει περισσότερο και με τη διαφορά κουλτούρας μεταξύ των δύο πλευρών. Ελπίζω όμως ότι και τα κρατικέ και οι κυβερνητικές οργανώσεις θα είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτή την συμφωνία προς όφελός τους. Η έκθεση δεν είναι ιδιαίτερα μακροσκελής. Για διάφορους λόγους. Βασικά ήθελα να είμαι συνοπτικός και ξεκάθαρος, όμως υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται σε αυτές τις εκθέσεις. Χαίρομαι λοιπόν ε, που τώρα πλέον μπορείτε να την διαβάσετε και στη συνέχεια με χαρά μου να απαντήσω σε ερωτήσεις, να γίνει συζήτηση, να γίνουν διορθώσεις εάν απαιτείτε. Να υπογραμμίσω επιπλέον ότι οι τροπολογίες πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Αν έχετε τροπολογίες, με χαρά μου να τις δεχτώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάνν Φέλτ. Δυστυχώς ε, πολλοί από τους σκιώδεις εισηγητές ε, δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μπούχνερ λοιπόν θα πάρει πρώτος το λόγο. Όχι, όχι, όχι. Ο Μάρτιν Φιρενσουστέρ πρώτος. Ναι. Ε, δεν ήταν εδώ, δεν είναι εδώ ο συνάδελφος, αλλά θα μπορούσα να διαβάσω ε, τη δήλωσή του. Ναι, δεν θα τα κατάφερνα έτσι κι αλλιώς. Λέει λοιπόν. Καλωσορίζω το γεγονό ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπολίου Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Κορέας έχει συμβάλει σε ε, την ε, βελτίωση ή στην ανατροπή μάλλον του ελλείμματος σε πλεόνασμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο κεφάλαιο 13.4 ε, η ε, ε, Κορέα έχει δεσμευτεί να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιό της έτσι ώστε να προβλέψει την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, την απαλυφή οποιασδήποτε μορφής υποχρεωτικής εργασίας, καθώς επίσης και την απαλυφή οποιασδήποτε διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά ε, την ε, απασχόληση, έτσι όπως ε, αναφέρονται και στη σύμβαση της Διεθνής, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Διαπιστώνουμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει σεβαστοί οι όροι της συνθήκης αυτής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε έχουμε δει ε, φυλάκιση διαμαρτυρώμενων εργαζόμενων ή συνδικαλιζομένων εργαζομένων οι οποίοι ζητούσαν ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ε, καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να προωθήσει τις ε, συγκεκριμένες μορφές ε, συμβάσεων. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι πολίτες μάλλον, δεν έχουν καλά ρυθμισμένη εργασία και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν οι διαμαρτυρίες ή οι, ή απεργίες να θεωρούνται παράνομες. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει επίσης ε, να ε, διαπιστώσουμε ότι είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες οι αρχές όσον αφορά την θέση, τη στάση των αρχών της Κορέας ε, απέναντι στους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους ε, και ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στην Κορέα όσον αφορά την, τις συνθήκες των εργαζομένων. Αυτά ήθελα να μας πει ο συνάδελφος. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι δεν μπορούμε να παρεύουμε στα εσωτερικά της Κορέας, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να προωθήσουμε τα εργασιακά ε, δικαιώματα και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ε, υπογραμμίσουμε πόσο σημαντικό είναι για μας η νέα κυβέρνηση να έχει καλές σχέσεις με τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους. Πρόεδρος, όντως Όντως η σχέση με τους ε, συνδικαλιστές δεν είναι πάρα πολύ ε, καλές μέχρι τώρα και επομένως ίσως ε, η συμφωνία να δώσει την ευκαιρία για μια καινούρια καλύτερη αρχή. Ο κύριος Μπούχνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σάνφελτ και τους συνεργάτες του για το σχέδιο αυτό έκθεσης, γιατί η έκθεση περιλαμβάνει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες και πολλά οικονομικά στοιχεία και είναι μια πολύ καλή αφετηρία για την περαιτέρω επεξεργασία μας και είναι δυνατόν να προσθέσουμε και τις δικές μας απόψεις με τροπολογίες. Εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ότι αυτή η πρώτη έκθεση εφαρμογής έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για περαιτέρω εκθέσεις αυτού του χαρακτήρα. Πρέπει να είναι λεπτομερής και εμπεριστατωμένη σε σχέση με το πώς έχει λειτουργήσει η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, επομένως να καταδείξει τις καλές και κακές πρακτικές και να προτείνει πώς μπορούν να βελτιωθούν. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της εποπτείας, το θέμα των εθνικών συμβουλευτικών ε, ε, επιτροπών και κυρίως το κεφάλαιο για την αηφορία. Εγώ ήμουν παρόν στην αντιπροσωπεία στη Νότια Κορέα που πήγε εφέτος και ένιωσα και κάποια έκπληξη για το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικά πορίσματα αυτής της επίσκεψής μας που δεν βρίσκονται στην έκθεση. Εν πάση νομίζω ότι είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει και μία αναφορά στις κέρυες αρχές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. <clears throat> Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές θετικές πλευρές σε αυτή την εμπορική συμφωνία. Θα πρέπει να δούμε την ε, αύξηση των εξαγωγών και τις, τους θετικούς μακροοικονομικές δείκτες. Η η αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών ουσιαστικά έγινε λόγω της ε, εξαγωγής αυτοκινήτων οχημάτων πολυτελείας, γερμανικών οχημάτων πολυτελείας προ τη Βόρεια Κορέα. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν θέλουμε μια εμπορική συμφωνία να ευνοεί μονάχα μερικέ ευρωπαϊκές εταιρείε και όχι τις δύο πλευρές εν γέννη. Εκφράζω την ικανοποίησή μου, εν για τη συνεργασία που είχα από τον εισηγητή και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και ξαφνικά είδα ότι οι Γερμανοί πράσινοι υποστηρίζουν τα γερμανικά οχήματα πολυτελείας. Καλά, αυτό είναι αστείο, λέει ο πρώτος, βέβαια. Δεν το εννοώ σοβαρά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος ζητά το λόγο και θα έλθω στην Κομισιόν. Φίλιπτε Μοντέι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για, την πολύ, για τα πολύ θετικά και χρήσιμα σχόλια που κάναμε σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι η έκθεση δείχνει ξεκάθαρα ότι η συμφωνία είναι μια συμφωνία επιτυχίας, ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από μια δεκαετία αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου με την Κορέα, έχουμε επιτύχει πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, έχουμε μια ολοκληρωμένη εξπόστα αξιολόγηση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βόρειας, Νότιας Κορέας που καλύπτει όλους τους τομείς. Η αξιολόγηση ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούλιο και ε, επιλέξαμε τον σύμβουλο ε, σε εκείνη τη φάση. Ελπίζουμε ότι τον Αύγουστο του 2017 θα έχουμε την τελική ε, έκθεση. Έχουμε και ένα link στην αρχική έκθεση στο site μας. Ε, επανερχόμενοι τώρα στην εφαρμογή. Οι τομείς που χρειάζονται περισσότερη επεξεργασία είναι ειδικά η, το SPS, δηλαδή έχουμε προβλήματα για το κρέας, το βόιο, αλλά και το ε, χοιρινό. Επίσης, ε, το IPR, ε, τα δικαιώματα δημοσίων ε, δημόσιας επίδοσης, επίσης ε, η κατάσταση των εργασιακών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Κορέα. Για την παρακολούθηση αυτής της εφαρμογής υπάρχουν αρκετές ομάδες εργασίας. Η Επιτροπή Εμπορίου στο επίπεδο της ε, Επιτρόπου Μάλστρομ θα συναντηθεί στις 16 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και έχουμε όσο περισσότερες συναντήσεις μπορούμε, ε, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πιο πριν. Έχουμε σε υπουργικό επίπεδο ε, συναντήσεις που θα συζητήσουν τα μεγάλα κεφάλαια. Παράλληλα, εξετάζουμε ειδικού τομείς της συμφωνίας για να δούμε πού ακριβώς βρίσκονται τα ωφέλη για τους εξαγωγείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ε, τροποποίησης της ε, συμφωνίας ε, τους όρους για τις άμεσες μεταφορές, όρους που έχουν να κάνουν με την αεροναυτική βιομηχανία, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα κεφάλαια τις, ε, που αφορούν στις επενδύσεις, ε, να ξέρετε ότι αυτή εδώ η συμφωνία ήταν πριν από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και δεν είχε συμπεριλάβει τις επενδύσεις. Όμως, έχει με τα κράτη-μέλη διμερείς συμφωνίες η Κορέα για αυτό το θέμα. Να πάμε τώρα σε δύο συγκεκριμένα θέματα, τα οποία νομίζω ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Καταρχάς, το κεφάλαιο εμπορίου και βιωσίμου ανάπτυξης. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά την κατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων στην Κορέα. Η συμφωνία προβλέπει έναν ε, θεσμικό μηχανισμό ε, σύμφωνα με τον οποίο τα μέρη συζητούν τα ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένων και των εργασιακών δικαιωμάτων, η Επιτροπή που συναντήθηκε πέρυσι στη Σεούλ ε, στην ουσία ε, είδε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητά από τη Σεούλ να επιταχύνει τα βήματα προς την ενίσχυση αυτού του τομέα. Στην κοινή δήλωση που εγκρίθηκε η Κορέα δεσμεύτηκε να παράσχει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα βήματα που προτίθεται να κάνει σε αυτή την κατεύθυνση πριν από την επόμενη συνάντηση της αντίστοιχης επιτροπής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να πιέζουμε σε αυτόν τον τομέα, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός για μας. Η Επιτροπή Εμπορίου θα λάβει χώρα στις 16 Δεκεμβρίου. Θα συμπροεδρεύει η Επίτροπος Μάλστρομ. Όσον αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, στις οποίες θέλουμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, διότι θα είναι και ξεκάθαρη δικαιούχη της συμφωνίας, κάνουμε το εξής. Η Επιτροπή δίνει πληροφορίες και εξειδικευμένα πρακτικά εργαλεία όπως μπροσούρες. Μέσω της ιστοσελίδας έχουμε και την βάση δεδομένων για την πρόταση στην αγορά που δίνει online δωρεάν πληροφορίες για τους δασμούς, την αγορά, τις απαιτήσει της αγοράς, στατιστικές, εμπορικές ροές κτλ. Έχουμε επίσης και το, ε, ε, την πύλη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων που δίνει πληροφορίες για την Κορέα και έχουμε και την πρωτοβουλία της, του δικτύου Enterprise Europe που έχει πάρα πολλούς εταίρους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες εκτός αυτής που μπορούν να υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της αγοράς της Κορέας. Επίσης βλέπουμε μια ξεκάθαρη αύξηση ε, των εξαγωγών στην Κορέα, 47%. Ε, νομίζω ότι αν ευαισθητοποιήσουμε για την ε, συμφωνία και μάθουν οι επιχειρήσεις, οι οργανώσεις και τα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνα για την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων θα μπορέσουν όλοι να εμπλακούν και να δώσουν τα σχετικά στοιχεία μέσα από τα εθνικά κανάλια μέσα από τα εμπορικά επιμελητήρια, για παράδειγμα, για να μπορέσουν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι εξαγωγές. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πιστεί πλήρως ότι η Επιτροπή πιέζει για τη σωστή εφαρμογή των κεφαλαίων για τη βιωσιμότητα σε μεγάλο βαθμό, γιατί εμείς έχουμε διαφορετική εμπειρία. Ξέρουμε ότι το Domestic Advisory Group δύο φορές ζήτησε να αναλυφθεί η δράση και η Κομισιόν δεν έκανε τίποτα. Και δεύτερον, υπάρχει μεγάλη ανάγκη αλλαγής. Πρέπει, λοιπόν, ε, να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ε, ειδικά στο ποινικό κομμάτι δεν γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι η Κομισιόν πιέζει για τη σωστή εφαρμογή του κεφαλαίου για τη βιωσιμότητα. Και κάθε φορά λέμε ότι θα γίνει άλλη μια συνάντηση, άλλη μια επιτροπή, αλλά μετά θα να θυμόμαστε ότι αυτή η συμφωνία είναι ακόμα σε δοκιμαστική φάση εδώ και πέντε χρόνια. Θα ήθελα πραγματικά μια πιο προμήθη και όχι επιμήθη επιτροπή. όσον αφορά τη στρατηγική για το εμπόριο. Αυτό ήταν δικό μου σχόλιο. Τώρα, να επανέλθουμε στον εισηγητή μας. Παρακαλώ. E, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής, ε, της δικής μας και τα μέλη της ε, ε, Κομισιόν, τους εκπροσώπους μάλλον της Κομισιόν που πήραν τον λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και σχολείων που δείχνουν ότι όλοι αποδίδουμε μεγάλη σημασία ε, στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε και εφαρμόζουμε τις συμφωνίες ελευθερού εμπορίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τις επιτηρούμε. Ε, είναι καλό να βλέπουμε και τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πλευρές ε, της υλοποίησης. Γιατί διαφορετικά δεν θα επιτύχουμε τους στόχους της συμφωνίας. Ε, στην περίπτωση των ε, συμφωνιών ε, ελευθέρου εμπορίου. Οπωσδήποτε, στην περίπτωση της Κορέας, θα γίνει λόγος σε επενδύσεις. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα πάμε καλά όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, ε, γιατί τα σχετικά κεφάλαια είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι απτά τα κριτήρια που χρησιμοποιούν. Όσον αφορά τώρα τα μη οικονομικά ζητήματα, αυτά τα οποία είναι ευθύνη κατά κάποιο τρόπο των δημοσίων αρχών. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Μιλείς μονούμε ότι εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετικές ε, ε, κουλτούρες. Μιλάμε για ε, πολιτισμό έτσι τελείως διαφορετικό. Άλλες είναι οι συνήθειες, ας πούμε, της ε, αγγλοσαξονικής αντιμετώπισης της εργασίας ε, και του ε, συνδικαλισμού. Διαφορετικά είναι τα πράγματα στην Ασία και στην Αφρική. Και Επομένως, όταν μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα, όταν μιλάμε για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, όταν μιλάμε για δικαίωμα ε, σε συνδικαλισμό κτλ., ε, η υλοποίηση αυτών των στοιχείων είναι πολύ πιο δύσκολη, διότι υπάρχουν ε, υπάρχουν πολιτιστικές και ε, ε, διαφορές, υπάρχουν εμπόδια τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη ζωή ε, οι άνθρωποι. Οπωσδήποτε όμως Πιστεύουμε ότι αυτές οι συμφωνίες FTAs μπορούν, ε, ελευθερού εμπορίου, ε, μπορούν να προωθήσουν ε, και αυτές τις αρχές. Και επομένως πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία και μια καλή επιτήρηση. Έχω ε, την αίσθηση πάντως ότι πολύ θετικά θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής μας ότι αυτή είναι η πρώτη έκθεση υλοποίησης και οπωσδήποτε εστιάζεται στην Νότια Κορέα, αλλά θα αποτελέσει ε, τον μορφότυπο, τον στάνταρ μορφότυπο ε, όσον αφορά τις ε, εκθέσεις υλοποίησης. Επομένως είναι μια μεγάλη ευθύνη που έχουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα καλό πρότυπο όσον αφορά τον έλεγχο της υλοποίησης και είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε το σαφές μήνυμα ότι η Επιτροπή μας δεν είναι μόνο υπεύθυνη για την διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών αλλά και για την υλοποίηση αυτών των ε, ε, συμφωνιών και επομένως ε, θα πρέπει να καλυφθεί και αυτό το σκέλος και επομένως ε, οι μελέτες υλοποίησης είναι και θα είναι πολύ σημαντικές. Ωραία ήταν η ευκαιρία λοιπόν, συζητήσαμε με τον εισηγητή και μέχρι την 9η Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε τροπολογίες. 9 Δεκεμβρίου 5 η ώρα το απόγευμα και ενδεχομένως στις 24 Ιανουαρίου θα γίνει και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Πολλή δουλειά λοιπόν έχουμε μπροστά μας αν θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή έκθεση υλοποίηση τη συμφωνία με την Νότια Κορέα, που θα αποτελέσει, είπαμε, και τον μπούσουλα για τα υπόλοιπα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, λοιπόν, η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 10, άρα μέχρι τότε τους ζυγούς λύσαμε. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Dann fangen wir mit den Abstimmungen an. Zunächst. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε. Καταρχάς, ε, θα ελέγξουμε λίγο τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Οπότε θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία καταρχήν. Ξεκινά λοιπόν η δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Όλα πάνε καλά, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάμε στο σημείο 12. Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κοινότητα ατομικής ενέργειας ε, όσον αφορά στο κοσυφοπαίδιο. Και εδώ έχουμε μια σειρά από τροπολογίες. Ξεκινάμε με την 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 13 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται η τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Και ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Συγγνώμη, δεν έχω την κάρτα μου. Μπορώ να ψηφίσω έτσι. Είμαι υπέρ. Και εγώ, γιατί η κάρτα μου δεν λειτουργεί. Ανάποδα νομίζω. Την βάζετε. So, vote by hand. So... Ωραία, ψηφίστε με διανατάσει τη χειρός. Δύο κατά. Όχι. Υπέρ. Ένας υπέρ και ένας κατά. Ωραία, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, 27 υπέρ, 2 κατά. Μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστούμε. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 13. Ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε περισσότερο είναι η προσχώρηση του Εκουαδόρ στην Συμφωνία Κολομβίας-Περού. Έχουμε μόνο μία ψηφοφορία και την κάνουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πού? Abstimmung ist geschlossen. Πέρας της ψηφοφορίας. Πώς θα ψηφίσετε ε, εσείς, παρακαλώ. Τώρα δούλεψε η κάρτα σας. Ωραία. Άρα μία επιπλέον ψήφος υπέρ, 25 υπέρ. Και πάλι με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, συγχαρητήρια στον κύριο Σόλτς. Ωραία. Αυτό ήταν ο γύρος των ψηφοφοριών, σύντομος και χωρίς κανένα πρόβλημα. Και πάμε τώρα Monitoring Gruppen. στις ομάδες παρακολούθησης. Monitoring Έχουμε δύο συναντήσεις που έγιναν πριν από την τελευταία, μετά την τελευταία συνεδρίαση. Ε, ε, το ένα ήταν Ασία, το άλλο τη Ασία μάλλον και το άλλο τίζα. Ειδικότερα το θέμα της, ε, το αιτήματος της Sri Lanka για το GSP Plus και είχαμε και τον πρέσβη της Sri Lanka που παρέστη. Η κυρία Καρυμλίπη, Δεν θα έχουμε κάποιον λοιπόν να μας πει σχετικά και μετά έγινε και στις 17 Νοεμβρίου μια ομάδα παρακολούθησης για την ΤΙΖΑ με τον κύριο Κίνερ, τον βασικό διαπραγματευτή. Είχαμε τον δεύτερο γύρο από τις 2 ε, μέχρι 10 Νοεμβρίου και είχαμε μια σειρά συζητήσεων. Φαίνεται όμως ότι στον τομέα αυτό η νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θέλει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, οπότε θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει, αν δηλαδή τελικά θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις ή όχι. Αυτό θα το δούμε με τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το επόμενο έτος, όταν πια ε, αναλάβει καθήκοντά της. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις, άρα πάμε στο σημείο 15. Η εισαγωγή ε, αυτόνομων μέτρων ε, εμπορίου για την Ουκρανία σύμφωνα με τη Συμφωνία Σύνδεσης προσωρινών μέτρων. Από την 1η Ιανουαρίου φέτος, όπως γνωρίζετε όλοι, είχαμε βαθιές και ολοκληρωμένες ε, συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας που προσωρινά χρησιμοποιούνται και εδώ αυτά τα έγγραφα στην ουσία μας μιλάνε για τις περαιτέρω παραχωρήσεις που θα υπάρξουν στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών. Έχουμε επίσης ε, τον, ήδη συζητήσει τον Οκτώβριο την εφαρμογή της συμφωνίας και έχουμε και στις ομάδες παρακολούθησης ε, μόνιμη παρακολούθηση. Σήμερα θα είναι η πρώτη συζήτηση για τις διευρυμένες αυτές προοπτικές. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον εισηγητή και χθε μας είπαν από την Κομισιόν ότι σήμερα θα μας δώσουν και αυτοί κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, η Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου με την Ουκρανία εφαρμόζεται προσωρινά από τον Ιανουάριο του 2016 η καθυστέρηση εφαρμογής οφείλεται στην πίεση της Ρωσίας. Αλλά ενδιαμέσως στις 29 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση για την εξαγωγή προσωρινών εμπορικών μέτρων στην Ουκρανία που συμπληρώνουν αυτά τα οποία θεσπίζονται βάσει συμφωνία σύνδεση. Τα μέτρα αυτά είναι ασυμμετρικά και έχουν σε στόχο να ενισχύσουν την Ουκρανική οικονομία και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες να γίνει μετάβαση σε μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς. Τα μέτρα αυτά θα σημαίνουν μηδενικούς δασμούς, ποσοστός μηδενικού δασμού για τα προϊόντα που είναι στα παρατήματα 1 και 2, επιπλέον των προτιμησιακών δασμών που προβλέπονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης, εν ε, μέρη πλήρη άρση τον ε, δασμό για προϊόντα της κατηγορίας του παρατήματος 3. Το παράτημα 1 και το παράτημα 2 περιλαμβάνουν αγροτικά προϊόντα όπως είναι το κρυθάρι, ο αραβόστος, το σιτάρι, το μέλι, ο χυμός, το χυμός σταφυλιού και οι ντομάτες και επίσης περιλαμβάνονται προϊόντα όπως είναι το αλουμίνιο, τα τρόφιμα, ηλεκτρικά μηχανήματα κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε και τα άρθρα για την ε, προσωρινή ε, διακοπή και μια ρήτρα διαφύλαξη σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά τα οποία θα εισαχθούν από την Ουκρανία θέσουν σε κίνδυνο ή δημιουργήσουν σοβαρέ δυσκολίε στου παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει να γίνουν περαιτέρω αξιολογήσει λόγω του γεγονότο ότι ο κανονισμό αυτό θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία του ταχύτερο δυνατό. Τα στοιχεία που έχουμε τώρα διαθέσιμα είναι μόνο από το 2007 πριν από την εφαρμογή τη συμφωνία ελευθέρων Εμπορίου. Γι' αυτό εγώ προσπαθώ για το θέμα αυτό να είμαι στο δυνατό πιο περιεκτικό. και άκουσα τι απόψει των εμπλεκομένων Ξέρω ότι η Επιτροπή Άγκρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζει μια γνωμοδότηση και θα ακούσω με προσοχή αυτά που έχουν να μπουν για τα προϊόντα αυτά. Γιατί ορισμένε διατάξει τη συμφωνία αυτή μπορούν να έχουν επιπτώσει σε ευαίσθητα προϊόντα των κρατών μελών. Γνωρίζω επίση ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγάλε προκλήσει αυτή τη στιγμή λόγω τη στρατιωτική αντιπαράθεση και τη απώλεια εδάφου και τι ιδιαίτερα πολυδάπανε μεταρρυθμίσει που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Πάνω τις ε, ε, ευρείες μεταρρυθμίσεις που γίνονται. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχάσουμε όλα αυτά, αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε μια ε, προτιμησιακή μεταχείριση σε εμπορικό επίπεδο. Προβλέπεται η ψηφοφορία για το θέμα αυτό να γίνει τον Μάρτιο στην Επιτροπή μας και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Αυτά είναι ρευστά, μπορεί να αλλάξουν γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες γνωμοδοτήσεις αλλά προς το παρόν αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Η Μέτα Ούτσκοκ δεν είναι παρούσα, αλλά μπορεί να μιλήσει ο Ντέβιτ Μάρτιν, εξ ονόματος. Θα διαβάσω μια δήλωση από την Μαρίτα Ούτσκοκ, όχι στα σουηδικά ευτυχώς. Ίσως τα σουηδικά είναι τα πιο απλά από τα γερμανικά, εν Λέει η Μαρίτα ότι η Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία, η οποία έτυχε διαπραγμάτευση το 2014, ήταν τελείω διαφορετική μακροοικονομική συγκυρία από αυτή που αντιμετωπίζει σήμερα η Ουκρανία. Αυτά ήταν πριν από την αρχή του πολέμου στον Τόνπα και την απώλεια εδάφους από, από τον έλεγχο της Ουκρανίας. Έχει υπάρξει κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο με τη Ρωσία που αυξάνει τις υποκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήδη δοκιμαζόμενη Ουκρανική οικονομία προτείνει η Κομισιόν να δώσει περαιτέρω αυτόνομες προτιμήσεις εμπορίου στην Ουκρανία για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθεί η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα αυτή. Αλλά τα έκτακτα αυτά, τα πρόσθετα μέτρα δεν μπορούν να είναι μια επιταγή λευκό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για του σοσιαλιστέ και δημοκράτε είναι απαραίτητο τα νέα αυτά αυτόνομα μέτρα να σέβονται τις ίδιες βασικές αρχές <clears throat> όπως αυτά που προβλέπονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης, δηλαδή σεβασμό για τις δημοκρατικές αρχές, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδης ελευθερίας και σεβασμός για την αρχή του κράτους δικαίου που είναι αδιαπραγμάτευτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η πρόταση Κομισιόν περιλαμβάνει και τέτοιες διατάξεις. Θα συνεχίσουμε επίση να τονίζουμε προ την Ουκρανία ότι πρέπει να κάνουμε πρόοδο σε θεσμικά θέματα και στον αγώνα κατά τη διαφθοράς. Πάνω απ' όλα θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι απλοί πολίτες, οι μικρομεσαίε ε, επιχείρησει να μην είναι στην υπηρεσία των ολιγαρχών. Αφλιώ όλα αυτά τα μέτρα δεν θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Θέλουμε επίση να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα εμπορικά μέτρα δεν θέτουν σε κίνδυνο ευαίσθητου ευρωπαϊκού οικονομικού κλάδου. Γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσουμε όλε αυτέ τι ποσοστώσει και τα πρόσθετα μέτρα προσεκτικά. Προσβλέπω στη συνεργασία με τον κύριο Βαλέσα και του άλλου οικειώδει. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ. Εκπρόσωπος του ΙΣΙΑΡ δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο Στέφαν Μπάλε δεν είναι εδώ. Ο κύριο Σούλτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ε, ο εισηγητής και ο Ντέιβιτ Μάρτιν ε, για τους ε, σκιώδεις και να σας πω ότι όταν συζητήσαμε το μικρό financial support πριν που είχαμε συζητήσει και πάντα λέγαμε ότι θα πρέπει να καλύπτει ε, και ε, τις κοινωνικές και οικονομικές ε, πτυχές. Αυτή ήταν σαφής προϋπόθεση και είχαμε πει τότε ότι είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί, διότι είχαμε την αίσθηση ότι η κατάσταση, και συμφωνώ με αυτά που ακούστηκαν, ε, είναι ήδη δύσκολη και επομένως ε, θα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο σε περίπτωση συμφωνίας σύνδεσης και πρόθεσης της. Ε, πώς να σας το πω. Δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η βοήθεια για τους στόχους που έχουν ε, δηλωθεί. Επομένως, η, λύπη ε, η διαφάνεια όσον αφορά αυτό το σκέλος της ε, βοήθειας. Χρειαζόμαστε επιπλέον διασφαλίσεις. Παρακολούθησα τη συζήτηση σχετικά με την τελευταία διάσκεψη κορυφής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Ε, γνωρίζουμε όλοι ότι ε, υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες των Υπουργών Εξωτερικών των σαν χωρών έτσι ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Βεβαίως πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση της Συμφωνίας του Μίνσκ ε, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα όμως ε, ακούμε και πολλά νέα σχετικά, από την Ουκρανία σχετικά με το κράτος δικαίου, σχετικά με βασικά ε, δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες για τους πολίτες. Επομένως, πολύ επικριτικά τα βλέπω όλα αυτά και περιμένω να δω τι θα γίνει και να προσπαθήσω βέβαια να καταλάβω και να έχουμε και πληροφορίες από την Κομισιόν για να δούμε ακριβώς που βρισκόμαστε, γιατί όλα αυτά συνδέονται και με το ε, ζήτημα ε, ας πούμε επισκεφτήκαμε επισκεφθήκαμε το ε, Κίεβο με τον διαμεσολαβητή και ξέρουμε ότι ε, και στο κέντρο της πόλης αλλά και στις ανατολικές της, ε, ε, της χώρας, συγγνώμη, και στις ανατολικές περιοχές υπάρχει ανάπτυξη οικονομική, επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται εκεί, επομένω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Χαουτάλα, τους πράσινους, ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι ακόμα μέλος, αλλά ελπίζω ότι θα γίνω σύντομα. Παρακολουθούμε και από τη Euronest πολύ στενά το θέμα αυτό. Βεβαίως η αρμόδια καθήλη είναι η Επιτροπή είναι και ε, ασχολείται με το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής της Ουκρανίας ήταν πάρα πολύ θετική, ε, διότι υπέφεραν πολύ από τα μέτρα που επέβαλε η ε, Ρωσία λόγω της προσέγγισης της χώρας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε θετικά ε, το θέμα της, του εμπορίου με την Ουκρανία. Υπάρχουν όμως ακόμα κάποια πραγματάκια που θα πρέπει να δούμε. Τα εμπορικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται, να ισχύουν και για την Κρυμαία και για τον Τόμπας. γιατί βεβαίως ε, ε, η Ουκρανία δεν αναγνωρίζει την ρωσική παρουσία και κατοχή σε αυτά τα εδάφη και επομένως αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερος. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο κατάλογος των προϊόντων τα οποία ε, ε, ενσωματώνονται σε αυτόν τον εμπορικό κατάλογο δεν αφορούν μονάχα μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να βοηθηθούν και οι μικρές επιχειρήσεις της ε, Ουκρανίας έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις ε, απασχόλησης. Ξέρετε ότι η ανεργία ειδικά των νέων είναι πολύ μεγάλη στην Ουκρανία. Πρέπει να το προσέξουμε και στις χώρες μας, αλλά αυτό η Ουκρανία μας απασχολεί τώρα. Ε, αυτό που είπε και ο συνάδελφος Μάρτιν και ο συνάδελφος Σόλτς προηγουμένως. Ε, ε, εάν δει κανείς το άρθρο 2 ε, της ε, πρότασης, προϋποθέσεις για την εφαρμογή των προτιμησιακών συμφωνιών και συνδέονται με το άρθρο 3 και την προσωρινή άρση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα αυτό, όπως το πρότεινε και ο Ντέιβιντ Μάρτιν, εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Χρειαζόμαστε ισχυρά μέτρα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχουμε διαπιστώσει κάποια πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα και δυσκολίες, ε, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πραγματικά ε, η νέα υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε το πώς, τον τρόπο με τον οποίο ε, θα διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της υπηρεσίας του Γενικού Εισαγγελέα αλλά και ε, ταυτόχρονα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει υψηλού προφίλ ε, πολιτικής υφής υποθέσεις διαφθοράς με ανεξάρτητο τόπο. Στο Κίεβο επίσης υπάρχει αυτή η συμβουλευτική αποστολή η οποία κάνει ε, πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι θα πρέπει να έρθω σε επαφή και με αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Η FTD. E Λυπάμαι που δεν είναι κανείς από την ομάδα του ECR γιατί για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Πάντα λένε ότι δεν είμαστε εδώ εμείς αλλά τώρα δεν είναι αυτοί εδώ. Εν πάση χρησιμοποιώ την ευκαιρία να Καλώς ορίσω την κυρία εδώ. Είναι πολύ καλό το να <clears throat> προσβλέπουμε στην παρουσία σας στην Επιτροπή μας και εγώ θα ήθελα να γίνετε μόνιμο μέλος από το τέλος του χρόνου όπως προβλέπετε. Θέλω επίσης να κάνω κάποιες ε, μακροπαρατηρήσεις. Εμείς υποστηρίζουμε βασικά το εμπόριο και λέμε εμπόριο και όχι βοήθεια. Αλλά ανησυχώ όταν οι εμπορικές συμφωνίες χρησιμοποιούνται ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Οι δικοί μου εκλογείς δεν θέλουν να πολεμήσουν με τη Ρωσία για την Κρυμαία, ούτε θέλουν οι εκλογείς μου να πολεμήσουν με τη Ρωσία λόγω της Ανατολικής Ουκρανίας. Και εδώ βλέπουμε κάποια ανησυχητικά δείγματα του ότι υποκρύπτεται κάτι πίσω από όλα αυτά και όχι απλώς η εισαγωγή ε, μελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εμένα μου αρέσει το μέλι βέβαια. Χαίρομαι για το φυσικό μέλι από, τις, από την Ουκρανία. Αυτό είναι θετικό αλλά θα ήθελα να σταθώ σε δύο μοναχα πρώτας και εδώ θα κλείσω. Λέει το κείμενο, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει και πάλι την στενή και πλήρη εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Πρώτη παράγραφος και η τέταρτη παράγραφος λέει η πρωτοβουλία αυτή της Κομισιόν θα πρέπει να ατενιστεί ως μια μορφή απτής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Η ομάδα μου λοιπόν και εγώ ανησυχούμε γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς την άρση των δασμολογικών φραγμών, των εμπορικών φραγμών, αλλά ότι αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη μορφή εξωτερικής πολιτικής <clears throat> και δεν νομίζω ότι έχει η Κομισιόν σκεφτεί τις ε, συνέπειες αυτής της πράξης. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. ENFF, ο κ. Όμπερ Μάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. οι απαιτήσει πλαίσιο για τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Όμως να μην απατώμαστε, ζητούνται πάρα πολλά, πράγματα που δεν έπρεπε να υπάρχουν ε, ε, είναι εκεί ε, δεν μπορούμε να δώσουμε μία λευκή επίταγη. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει το κράτος ε, δικαίου. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο και ούτε καθεξής. Ε, η κατάσταση αυτή τη στιγμή φαίνεται τελείως διαφορετική. Βλέπουμε αποχωρήσεις υπουργών που είχαν άλλες προσδοκίες πάνω ας πούμε στο εξωτερικό στη Γεωργία και σε αυτήν εδώ την έκθεση βλέπουμε ότι είναι κάπως διπλωματική θα πρέπει κανείς, αν τα δει όλα με ησυχία, να καταλάβει ότι χρειάζεται να πάμε εκεί. Η αντιπροσωπεία στην Ουκρανία είχε κάνει πολύ καλές ε, συζητήσεις και δεν βλέπουμε καμία πρόοδο σε επίπεδο κράτους δικαίου. Υπήρξε μία ε, ε, φιλόδοξη επιστολή για την διαφθορά και την πάταξη της διαφθοράς όμως δυστυχώς ε, βλέπουμε ανθρώπους που μπαίνουν στην ε, φυλακή και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και δεν ε, απονέμεται η δικαιοσύνη όπως πρέπει. Γενικά φαίνεται ότι όλο το σύστημα είναι διεφθαρμένο, έχουν ε, υπάρξει αστυνομικοί που έχουν εμπλακεί σε όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να αξιολογήσει τους όρους, ξεκάθαρους όρους, τους οποίους όμως μετά θα ελέγχουμε, θα τους τηρούμε και δεν θα λέμε πάντοτε το ίδιο, δεν θα δεχόμαστε τα πάντα, θα απαιτούμε αυτό που πρέπει να γίνει. Και αυτό για την δική μου ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Όταν υπάρχουν όροι, ειδικά για το κράτος δικαίου, δεν είναι διαπραγματεύσιμοι. Γιατί χωρίς αυτούς δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα να κάνω που καθαρίστηκε με τις συζητήσεις στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα λοιπάσματα τα οποία ε, ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τηρούνται. Πρόκειται για συγκεκριμένα συστατικά των δραστικών ουσιών και αυτό έχει να κάνει με την τοπική γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να το σκεφτούμε λίγο αυτό, το dual use, ε, διότι όταν ε, βλέπουμε παρόλο που υπάρχει η ακεχηρία, να έρχονται ολόκληρα ε, τρένα από την Ρωσία με πολεμοφόδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, μπορεί στην ουσία να τιμωρούμε την γεωργία και να μην έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τώρα ο κύριος Σουμίλης από την Κομισιόν. Yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολλά τα σχόλια, Απλώ θα ήθελα να σα δώσω ένα γενικό πλαίσιο, κάποιε βασικέ πληροφορίε σε σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν. Η πρόταση αυτή τη Κομισιόν έχει προετοιμαστεί λαμβάνοντα υπόψη τι πολύ στενέ σχέσει που έχουμε με την Ουκρανία μέσω τη συμφωνία σύνδεση και με την δημιουργία μια πλήρου περιοχή ελευθερών εμπορίου. Λαμβάνει φυσικά υπόψη την τωρινή πολύ δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία όχι μονάχα λόγω των περιοριστικών μέτρων και των ε, κυρώσεων που έχουν ε, υιοθετηθεί από τη Ρωσία όπως είπανε πολλοί από εσά. <clears throat> και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Ρωσία ήταν στο παρελθόν η κύρια εξαγωγική αγορά για την Ουκρανία, κάτι το οποίο τώρα έχει συρρυκνωθεί και έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η κύρια εξαγωγική αγορά για την Ουκρανία. Η πρόταση αυτή λαμβάνει υπόψη εξάλλου και τις προσπάθειες που έγιναν από τις Ουκρανικές αρχές για να εισαγάγουν μία σειρά από μεταρρυθμίσεις. Φυσικά είναι τιτάνια οι πρόκληση που αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά έχουν ήδη λάβει πολλά μέτρα και επίσης αυτό περιλαμβάνει και τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Την προηγούμενη εβδομάδα όπως ξέρετε, η διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας στις Βρυξέλλες και απετίμησε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις Ουκρανικές αρχές. Αυτό λοιπόν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Κομισιόν θεώρησε ότι ήταν σημαντικό να παρουσιάσει μια πρόταση για αυτόνομα εμπορικά μέτρα έναντι της Ουκρανίας που όπως είπε και κάποιο από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι ένα δείγμα απτής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Προετοιμάζοντας τώρα αυτή την πρόταση, η Κομισιόν ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και επέλεξε μια σειρά προϊόντων που είναι το αντικείμενο της πρότασης αυτής για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως ξέρετε έχει δύο πτυχές η πρόταση αυτή. Αφενός αφορά μια σειρά από γεωργικά προϊόντα αλλά επίσης έχει να κάνει και με ποιημένα βιομηχανικά προϊόντα. Για τα βιομηχανικά προϊόντα η Συμφωνία Πλήρους Ελευθέρου Εμπορίου είχε ήδη φιλελευθερωποιήσει το εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων. Επομένως υπάρχει μόνο ένα μικρό, μικρός αριθμός προϊόντων που υπόκειται σε μεταβατικά μέτρα και η πρότασή μας θέλει ένα γνήσιο υποσύνολο αυτών των προϊόντων που υπόκειται σε μεταβατική περίοδο να έχουν μικρότερη μεταβατική περίοδο. να έρθουν λοιπόν πιο σύντομα τα ε, περιοριστικά μέτρα για αυτά τα προϊόντα. Αυτό κάνουμε για τα βιομηχανικά προϊόντα. Για τα αγροτικά προϊόντα όμως, το εμπόριο με την Ουκρανία είναι σε μεγάλο βαθμό μέσω της Συμφωνίας Ελευθερου Εμπορίου φιλελευθερωποιημένα, αλλά υπάρχουν 36 προϊόντα που υπόκειται σε δασμούς από τα 36 αγροτικά προϊόντα που υπόκειται σε ποσοστό και δασμούς. Έχουμε επιλέξει 8 και για αυτά τα 8 προϊόντα προτείνουμε να διευρύνουμε το μέγεθος των ποσοστώσεων που θα μπορούσε να εξάγει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς πρόσθετους δασμούς, χωρίς δασμούς. Για τα περισσότερα από αυτά τα 8 προϊόντα η Ουκρανία εξάγει σημαντικές <clears throat> ποσότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνονται στις πρόσθετες ποσότητες που εμείς θα προτείνουμε με αυτή την πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι η πρότασή μας θα εξασφαλίσει την νομική ασφάλεια για τους εξαγωγείς από την Ουκρανία και θα σημαίνει ότι δεν θα χρειάζονται οι εξαγωγείς να πληρώνουν δασμούς για τις πρόσθετες αυτές ποσότητες αλλά αυτά τα προϊόντα ήδη εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και η επιλογή αυτών των 8 αγροτικών προϊόντων από τα 36 έγινε με τρόπο ώστε να αποφύγουμε να συμπεριλάβουμε προϊόντα τα οποία ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα. Τα, τα γαλακτοκομικά δεν είναι εκεί, το, τα πουλερικά και το κρέας δεν είναι μεταξύ των προϊόντων αυτών, γιατί όλα αυτά τα προϊόντα είναι ευαίσθητα, αλλά επίσης ε, <clears throat> περιλαμβάνονται και στις ρωσικές ε, ε, κυρώσεις κατά των εξαγωγών μας. Κάναμε λοιπόν μεγάλη προσπάθεια και με εργόδεις προσπάθειες έχουμε σταθμίσει σωστά την πρότασή μας και όπως ανέφερα και διάφοροι βουλευτές υπάρχει και μια διαδικασία <clears throat> διαφύλαξης και ένα άρθρο που περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρωθούν ώστε η Ουκρανία να υποφεληθεί από αυτά τα αυτόνομα μέτρα και πρόκειται για την συμμόρφωση με βασικές αρχές της πολιτικής ε, μπορεί όπως είναι οι κανόνες προέλευσης αλλά και η συμμόρφωση με γενικότερες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με το σεβασμό των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τελευταίο στοιχείο της πρότασης αυτής είναι ότι έχει ένα προσωρινό χαρακτήρα. Προτείνουμε λοιπόν να εφαρμοστεί όχι παραπάνω από τρία χρόνια, μόνο για μια χρονική διάρκεια τριών ετών και η περιορισμένη αυτή διάρκεια των τριών ετών σημαίνει για μας ότι από την οπτική γωνία της Κομισιόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να εγκριθεί ταχαίως το μέτρο αυτό γιατί αν είναι μονάχα για τρία χρόνια δεν πρέπει να καθυστερήσουμε την εφαρμογή του μέτρου αυτού και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να υποφεληθεί του μέτρου αυτού το ταχύτερο δυνατό. Γι' αυτό έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και έναντι του Συμβουλίου ζητούμε να υπάρξει μια ταχεία έγκριση αυτή τη απόφαση. Εάν υπάρχουν τώρα κάποια ερωτήματα που θέλουν τυχόν να θέσουν τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα διάφορα προϊόντα που εμπλέκονται, στην πρόταση της Κομισιόν <clears throat> δεν υπήρξαν ειδικέ ε, παρατηρήσεις για προϊόντα σήμερα, αλλά είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να δώσουμε τις πληροφορίες αυτές, είτε με τη μέρα, είτε εγγράφος, όπως θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Τι γίνεται με το κοτόπουλο και τμήματα ε, κοτόπουλου, καλύπτεται. Πολύ ωραίο, κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλους σας ευχαριστώ που συμμετείχατε σε αυτή τη σημερινή συζήτηση. Ε, και εδώ να συνοψίσω λίγο. Νομίζω ότι όλοι ε, έχουμε τις ίδιες κεντρικές ανησυχίες και έχουμε, συμμεριζόμαστε κατά κάποιο τρόπο τις ίδιες ε, κεντρικές ιδέες. Στην ουσία λοιπόν, δημοκρατικό κράτος δικαίου, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνέχιση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, πρόθεση της διαφάνειας, όπως είπε ο κ. Σόλτς, πολύ σημαντικό, συνδικαλιστική ελευθερία, ε, όλα αυτά τα μέτρα ε, δεν ε, θα πρέπει να υλοποιηθούν γιατί εμείς δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Πρέπει να εφαρμόσουμε και τις αρχές μας και πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία θεωρούνται βασικά στοιχεία ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, λέμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν όσο γίνεται ε, πιο γρήγορα αλλά πραγματικά θα πρέπει να έχουμε λίγο χρόνο έτσι ώστε να αναλύσουμε όλα τα μέτρα πολυεπίπεδα θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι εδώ, ε, τι είδους επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, στις διατάξεις, τι θα γίνει με τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, με την Κρυμαία. Η Κρυμαία αναφέρθηκε επίσης. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής κατά πόσον ε, οι διατάξεις ε, προωθούν ε, τις και βοηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα το μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα. Εν τέλει πιστεύω ότι όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πόρη, η μείωση των ποσοστώσεων και των δασμών δεν θα πάνε στράφη είτε μέσω κακής χρήσης, είτε ε, με λόγω ελλειπούς ε, υλοποίησης. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι και στην Ουκρανία εφαρμόζονται οι σύγχρονες ε, αρχές διασφάλισης έτσι, της υλοποίησης. Τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, το εμπόριο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ε, είναι εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το επιχείρημα ή από αυτήν την ε, κατηγορία, αν θέλετε. Έτσι είναι δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ για την ε, συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ισηγητά. Ο κύριος Σόλτ θέλει να υποβάλει ένα ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ κύριε Βαλέσσα. έχουμε συζητήσει ίδιες πτυχές, τα ίδια ερωτήματα πριν από δύο χρόνια, αλλά και πέρσι. <clears throat> Υπάρχουν ακόμα ολιγαρχικές δομές στην Ουκρανία. Βέβαια, αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάμε για εξειδίκευση κατά περιοχές. Αν δείτε όμως την ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επιβιώσουν, μπορούν με τη μακροοικονομική μας βοήθεια και τα άλλα μέτρα τα οποία προτείνουμε να αποσυνδεθούν και να είναι ανεξάρτητες από τις ολιγαρχικές αυτές δομές. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν σε ποιο βαθμό η βοήθειά μας συμβάλλει στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στην έκθεση να συμβάλλουμε για το θέμα αυτό αλλά θα ήθελα ίσως να μας δώσει και η Κομισιόν κάποια περισσότερη πληροφόρηση και γι' αυτό αναφέρθηκα και με την διαμεσολαβήτρια που ασχολείται για την ειδική κατάσταση των ε, μικρομεσαίων επιχείρησεων στην οικονομία και ξέρουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα παραγωγής από ολιγαρχικές δομές και τη Ρωσική Ομοσπονδία που διοχετεύεται στη χώρα. Λοιπόν, η κατάσταση της οικονομίας ακόμα δεν έχει την απαραίτητη διαφάνεια <clears throat> και γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουμε αυτό γιατί σε τελική ανάλυση <clears throat> οι εργαζόμενοι στους οικονομικούς κλάδους της Ουκρανίας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν, να βγάλουν το ψωμί τους με την εργασία τους και αυτό δεν είναι ακόμα προφανές, ιδίως στο κεντροανατολικό κομμάτι της ε, Ουκρανίας. Ο Μάιλ με χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση προς την Κομισιόν. Είναι γνωστό ότι υπάρχει παραγωγή ξύλου η οποία ε, έχει εμποδιστεί τώρα αυτή τη στιγμή και αυτό επηρεάζει και την ευρωπαϊκή βιομηχανία χαρτομάζας που βασίζεται στην ε, χρήση ξύλου από την Ουκρανία. Αν μπορεί να μας απαντήσει εσείς με το θέμα αυτό η Κομισιόν. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, να έρθω σε αυτό το θέμα του πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ουκρανία και για τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης ανασυγκρότηση για, την επένδυση, για τις επενδύσεις στη χώρα. Να διασφαλίσουμε ότι οι νόμοι για τις δημόσιες συμβάσεις διασφαλίζουν τη διαφάνεια και ότι οι διαγωνισμοί γίνονται σωστά. Υπάρχει ε, πολλή δουλειά ακόμα για, που πρέπει να γίνει στην Ουκρανία, καθώς ε, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία ε, ως προς τις διάφορες θετικές δυνάμεις που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία. Θα ήθελα να ακούσω και την Κομισιόν τι έχει να πει για τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Κομισιόν λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτή η συμφωνία με την Ουκρανία είναι το όχημα προς την μεταρρύθμιση. Αυτό είναι το πνεύμα της σημαντικές μεταρρυθμίσεις προβλέπονται για σημαντικούς ε, τομείς όπως ε, ας πούμε την γεωργία, δημόσιες συμβάσεις, υγειονομικά και φυτο μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα και τις στρατηγικές δηλαδή που αναπτύσσονται σε συνεργασία με την Ουκρανία. Κάποια από αυτά, ειδικά στον τομέα των δημοσίων ε, συμβάσεων, έχουν μεγάλη πρόοδο, Επίση, στα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα. Πάει πολύ καλά το πράγμα. Έχει ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση για τη στρατηγική. Λαμβάνουν χώρα λοιπόν πολλέ μεταρρυθμίσει ήδη. Επίσης, παρέχουμε συνδρομή διότι αν ε, στην ουσία αυτοί πρέπει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις να συμμορφωθούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που διαφέρουν από αυτά που ήδη υπάρχουν στη χώρα τους, ε, ε, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν την τεχνογνωσία, θα χρειαστεί κάποιες φορές να προσαρμόσουν τις επενδύσεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα τους τα οποία θα συμμορφώνονται με τα πιο αυστηρά στάνταρ. Και γι' αυτό έχουμε και διάφορα εργαλεία συνδρομής και βοήθειας. Αναφέρθηκαν πολλοί ευρωβουλευτές στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη διευκόλυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη λειτουργεί και λειτουργεί και μέσα από την παρέμβαση διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης ε, που ήδη αναφέρθηκε και άλλες. Το θέμα τώρα όμως είναι πώς συνδέουμε την αρρωγή, τη βοήθεια μέσα ε, με το εργαλείο που έχουμε στην πρόταση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με ένα γεωργικό προϊόν, το μέλι. Το μέλι είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι πολύ συγκεντρωμένο. Η παραγωγή του δεν είναι πολύ συγκεντρωμένη. Είναι κυρίως μικρές επιχειρήσεις, μικροί γεωργοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν το προϊόν. Όμως, μέσα από αυτό το εργαλείο, μέσα από τη διευκόλυνση, θα τους βοηθήσουμε να έρθουν στην αγορά μας. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχουν και άλλα. Απλώς για τη σημερινή συζήτηση σας ε, δίνω αυτό το παράδειγμα. Τώρα υπήρξε μια ερώτηση για τους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ουκρανία για το ακατέργαστο ξύλο. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και ένα χρόνο από τότε που η Ράντα έχει υιοθετήσει αυτή τη διάταξη για τις εξαγωγές. Το έχουμε θέσει σε όλα τα επίπεδα. Είναι και μία από τις αρεσιμότητες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ήδη γίνεται κάτι, υπάρχει κάποια πρόοδος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε επεξεργασία το σχέδιο της νομοθεσίας σχετικά με την άρση αυτής της απαγόρευσης. Την περασμένη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής έγινε αυτή η συζήτηση, υπήρξε μια μεγάλη περίοδος κατά την οποία επιμέναμε ότι αυτό το πράγμα ενοχλεί ιδιαίτερα ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διατάξεις της συμφωνίας μας. Τώρα βλέπουμε κάποια πρόοδο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η νομοθεσία που έχουμε συζητήσει έτσι δοκιμαστικά ε, θα μπορέσει σύντομα να εγκριθεί για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε το σχέδιο της έκθεσης στις 23 ή 24 Ιανουαρίου και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για όλη αυτή την άσκηση. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι τώρα πρέπει να πάμε στο, στην αίθουσα Γιάν 4Q1. Τέταρτος όροφος, το Q1 στο κτίριο Γιάν. Ξεκινάμε στις 11 την κοινή συζήτηση σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα στις συμφωνίες εμπορίου μαζί με την, ε, δηλαδή με την Επιτροπή Απασχόλησης. Στις 12.30 εδώ σε αυτή την αίθουσα θα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια για τη ΣΕΤΑ και στις 3 θα ξεκινήσουμε εδώ την κανονική μας συνεδρίαση ως συνήθως. David. Μια ερώτηση. 12 και ε, ε, υπάρχει μία, είναι ανοιχτή η συζήτηση μόνο για τα μέλη. Δεν είναι κλειστή, αλλά θέλουμε να γίνει συζήτηση μεταξύ των ε, μελών. Ε, δεν θέλω να πω ότι... Α, πάντως μεταξύ μελών.